Uh, Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ε, κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη ψηλού επίπεδου για την ανάπτυξη και την ε, μετανάστευση που είναι κοινή ε, δουλειά του ΟΣΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. χαιρετώ τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ σας καλωσορίζω το θέμα που μας ε, φέρνει σήμερα εδώ είναι πολύ σημαντικό σήμερα όλοι το ξέρουμε όλοι ξέρουμε την, την τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζουμε οι μετανάστες είναι 3% του ε, παγκόσμιου πληθυσμού 200 εκατομμύρια ε, άνθρωποι οι μετανάστες είναι ο τρίτος κατά σειρά μεγαλύτερος πληθυσμός η μεγαλύτερη χώρα θα ήταν αν ζούσαν σε μια χώρα σε ορισμένες χώρες βέβαια ενώ ο μέσος όρος είναι 30% τα, ε, η μετανάστευση έχει φτάσει στα 9-10% σε ορισμένες άλλες χώρες όπως την Ισπανία παραδείγματος χάρη το 20% αλλά η κινητικότητα είναι είναι ε, μεγάλη στην εποχή μας και γι' αυτό η, ε, οτιδήποτε σχετίζεται με την μετανάστευση έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, και στην Ευρώπη και αλλού. Είναι σημαντικό και οι κοινοβουλευτικοί να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και μετανάστευσης και σήμερα γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ όχι μόνο κοινοβουλευτικοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του κόσμου. Θα συζητήσουμε ε, δύο πολύ σοβαρά θέματα τα οποία τα χωρίσαμε σε δύο πάνελς που θα λάβουν χώρα σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο πάνελ για την ανάπτυξη και τη μετανάστευση και δεύτερο πάνελ για τις αγορές εργασίας, εργασίας και πώς ε, μπορούμε να διαχειριστούμε τη μετανάστευση και σε συνδυασμό με τις αγορές εργασίας που τόσο ώστε να, αυτό να ικανοποιεί τους πάντες. Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω εδώ σήμερα τον κύριο Πέτερινγκ πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κυρία Βάλστρομ την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Βάλστρομ είναι υπεύθυνη ε, για θέματα για τη σχέση μεταξύ των οργάνων στη, και για την επικοινωνία και το χαιρετώ επίσης και τον κύριο Αμάνο που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Λουί Μισελ που απρόκειτο να έρθει σήμερα δυστυχώς δεν μπορούσε να παραστεί διότι ασθενή έχει γρήπη ακόμη και επίτροποι παθαίνουν γρήπη που και που το ευχόμαστε ε, περαστικά και γι' αυτό στη θέση του ανακαλωσορίζουμε εδώ τον Αντιπρόεδρο αλλά πριν να αρχίσουμε τις συζητήσεις και τις ομιλίες ε, να κάνω μερικές πρακτικές παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα διερμηνία 20 22 γλώσσες υπάρχει διερμηνία ε, λείπουν τρεις γλώσσες αλλά νομίζω ότι είμαστε εντάξει θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε δεύτερον θα μοιραστεί σε όλα τα μέλη μία, ε, ένα έντυπο ε, για εγγραφής και θα θέλαμε να δώσετε τα στοιχεία σας ε, γιατί αυτό από εκεί και πέρα ε, ο χρόνος ομιλίας θα είναι περίπου δύο λεπτά και θα θέλαμε να τον τηρήσετε. Ε, το διάλειμμα το μεσημεριανό θα είναι από τις 12.30 μέχρι τις 2. Ε, έχουμε, θα διοργανωθεί ένας μπουφές μπροστά στην αίθουσα αυτή στην οποία, στον οποίο σας καλούμε όλους όλα μαγνητοσκοπούνται και βγαίνουν και από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταδίδονται σε όλες τις γλώσσες της ε, Ευρώπης live. Λοιπόν, Αυτά εισαγωγικά με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τον κύριο Πέτερινγκ. Σας ευχαριστώ με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ υπό την προεδρία του, του Γιώζεφ Μπορέλ όταν ο κύριος Μπορέλ ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγώ ήμουν πρόεδρος μιας πολιτικής ομάδας χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι εδώ ε, και τώρα θα συνεχίσω στα γερμανικά που είναι η μητρική μου γλώσσα κυρία Επίτροπε Βάλστρομ κυρία γενική Γραμματέα γιατί του όσα, κύριε Μάριο Αμάνο, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας καλωσορίζουμε εδώ με την ευκαιρία της σημερινής συνδιάσκεψης. Στόχος της σημερινής συνδιάσκεψης είναι να συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε στην ανάπτυξη και κυρίως στη μετανάστευση, στις πολιτικές μετανάστευσης των διαφόρων χωρών σε συνεργασία με τις, αναπτυσ... με τις τρίτες και αναπτυσσόμενες χώρες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία στενής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων απανταχού στον κόσμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει πάσα προσπάθεια ούτως ώστε να έχει στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Ο Γιώζεφ Πορέλ ε, ξεκίνησε την ιδέα αυτή επί προεδρίας του. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και εγώ και πριν από μερικές μέρες ήμουνα στη Φινλανδία για να συνεργαστώ ακριβώς με τους Φινλανδούς βουλευτές. Ως κοινοβουλευτικοί θεωρούμε ότι έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη για τους πολίτες μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα ήρεμο και ειρηνικό μέλλον παντού και για όλους μας. Η η συνέργεια μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Η, η μετανάστευση θα μπορούσε να είναι εργαλείο για ανάπτυξη, αγαπητοί φίλοι και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πολλές ε, πρωτοβουλίες σχετικά και όσα επίσης. Έχουν γίνει πολλές μελέτες και αναλύσεις για την ε, μετανάστευση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι πολιτικές των κρατών να έχουν, ε, να έχουν μια κάποια συνοχή, να είναι κάπου συντονισμένες ούτως ώστε να μπορούν τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ιδιαίτερα στις εθνικές κυβερνήσεις τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει σχετικά από εκεί και πέρα ελπίζουμε να φτάσουμε κάποια σε μια στιγμή όπου όλοι σε όλα τα πολιτικά βήματα ε, σε όλο τον κόσμο θα μιλούμε με μια φωνή για τα θέματα ανάπτυξης και μετανάστευσης. Η πολιτικές μετανάστευσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις πέρα από τις πολιτικές τους επιπτώσεις έχουν επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων αυτών που είναι μετανάστες και όπως ελέγχθη οι μετανάστες είναι η, ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός <coughs> μετανάστης γίνεται κανείς ε, είτε λόγω τεράστιας φτώχειας, λόγω προβλημάτων ε, θρησκευτικών, πολιτικών, πολιτικών σειράξεων, πολέμων ή οικονομικών προβλημάτων. οι μετα, λοιπόν μπορεί να γίνει κανείς για χίλιους δυο λόγους και γι' αυτό η μετανάστευση βρίσκεται στην ημερησία διάταξη όλων σχεδόν των πολιτικών όλων αυτών που ασχολούνται με την πολιτική. Η μετανάστευση επηρεάζει λοιπόν την ανάπτυξη αλλά και η ανάπτυξη επηρεάζει τη μετανάστευση. Η, τα αίτια και οι επιπτώσεις της μετανάστευσης ε, έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν και έχουν τονιστεί ιδιαίτερα κάποιες αρνητικές πτυχές της μετανάστευσης. Σήμερα θα δούμε τις θετικές επιπτώσεις γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι ο μετανάστης που φεύγει από μια αναπτυσσόμενη χώρα και επιστρέφει μετά στη χώρα του μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας αυτής επιστρέφουν άτομα με νέες γνώσεις με νέες ικανότητες με νέα προσόντα από εκεί και πέρα οι οργανώσεις της διασποράς μπορούν να συμβάλλουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις των χωρών προέλευσης και των χωρών υποδοχής. Αν ε, ε δεν ε, συμβούν αυτά που έλεγα προηγούμενα δεν επιστρέψει κάποιος με επιπλέον γνώσεις ας πούμε στη χώρα από την οποία ήρθε τότε ε, τα προβλήματα η, το, τότε οι επιπτώσεις μετανάστευσης είναι αρνητικές διότι συμβαίνει αυτό που ονομάζουμε brain drain φυγή εγκεφάλων από κάποιες χώρες πάνω από 55% των Νιγηριανών 39% των ε, από την ε, Ζαμπία, από το Λεσόθο, από την Ναμίμπια, από την Τανζανία και από την Νότια Αφρική ε, ε δουλεύουν εκτός των χωρών τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υψηλά προσόντα, υψηλές γνώσεις με, και έχουν καλές θέσεις εργασίας αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό 60% όλων των γιατρών που εκπαιδεύτηκαν στη Γάνα, Γάνα δουλεύουν στον Καναδά στις Ηνωμένε Πολιτείες και λιγότερο από 10% των γιατρών που εκπαιδεύτηκαν στη Ζάμπια μένουν και ασκούν το επάγγελμά τους στη χώρα τους. Είναι λοιπόν σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Είναι μια πρόκληση πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και τις αρνητικές πτυχές της μετανάστευσης η, σαν και αυτές που ανέφερα οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες φεύγουν οι εκπαιδευμένοι γιατροί ή οποιοδήποτε άλλοι επιστήμονες Κυρίες και κύριοι, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε ότι η μετανάστευση και στις χώρες μας και στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες προέλευσης είναι, έχει θετικές ε, επιπτώσεις για το θέμα της φτώχειας θα πρέπει να βρούμε εργαλεία και μέσα για να αντιμετωπίσουμε και εκεί τα σχετικά προβλήματα και η συνεργασία με τα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ έχει σαν στόχο να συντονίσει καλύτερα τα πράγματα Υπά, από το Δεκέμβριο του 2005 βεβαίως υπάρχει συνένεση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική ανάπτυξη, την αναπτυξιακή πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και η, η ευρωπαϊκή στόχη της, ε, στον τομέα της ανάπτυξης που ε, άπτονται και των αναπτυσσομένων χωρών θα πρέπει να ε, λαμβάνουν υπόψη και την ε, το φαινόμενο της μετανάστευσης και πραγματικά η μετανάστευση είναι ένα πολύ ε, σημαντικό θέμα και πολιτικές των μετανάστευσης των διαφόρων χωρών όπως είπα και πριν θα πρέπει να κάποια συνοχή, ένα κάποιο συντονισμό. Η... Οι εθνικές πολιτικές, άμα είναι συνεκτικές και ε, συντονισμένες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας που έχουμε αποφασίσει όλοι και βεβαίως θα πρέπει να συμμετέχουν στην ε, κατάρτιση των πολιτικών αυτών και όλοι οι ενδιαφερόμενες ομάδες, οι ομάδες στόχοι που εμπλέκονται στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Κλείνοντας κυρίες και κύριοι να πω ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις αλλά οι καλύτερες λύσεις βρίσκονται με συνεργασία και διάλογο και ο διάλογος αυτός θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εμείς εδώ η συνδιάσκεψή μας η υψηλού επίπεδου είναι ένα βήμα σε αυτό, στο διάλογο που πρέπει να γίνει μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. Ελπίζω ε, η σημερινή συνδιάσκεψη να μας ε, βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη συνειδητοποίηση και κατανόηση των φαινομένων με τα οποία ασχολούμεθα και θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις χώρες και θα ήθελα συνάδελφοι και φίλοι να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καρποφόρες συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και ευχαριστούμε και όλους αυτούς που δούλεψαν για τη διοργάνωση της ε, σημερινής συνδιάσκεψης. Thank you, President Muchas gracias, querido Hans ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Έχω την ευχαρίστηση να πάρω το λόγο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βάλστρουμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέμπλ, ε, αξιότιμα μέλη, Πρόεδρε κύριε Πέτερινγκ, μέλη του πάνελ. Είναι μια τιμή για μένα που έχω αυτή τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε μια τόσο διακεκριμένη συνδιάσκεψη που έχει τόσο πολλούς συμμετέχοντες από ολόκληρο το κόσμο. Και ε, ο συνάδελφος Λουί Μισελ λυπάται πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω και ταυτόχρονα θα ήθελε να σας ευχηθεί καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μου δώσατε το λόγο. Η συνεργασία και ο συντονισμός μοιάζουν φυσικά στοιχεία όταν υπάρχει ομαδική εργασία. Και αυτό λυθεύει ιδιαίτερα όσον αφορά την χάραξη δημόσιων πολιτικών, ούτω ώστε η μία πολιτική να μην επηρεάζει αρνητικά τι εφαρμογέ των άλλων πολιτικών. Ωστόσο προποθέτει ε, μια ιδιαίτερη σύνεση, είναι ε, μια ευαίσθητη διαδικασία εξισορρόπησης διάφορων ε, στοιχείων. Και αυτό και εδώ θα πρέπει ακριβώς αυτή τη συνεκτική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεκτική πολιτική της ανάπτυξης είναι ε, ο άξονας αυτός, το μοντέλο το οποίο βοηθάει να εξωσορροπήσουμε αυτά τα στοιχεία. 12 ε, επιλεγείς πολιτικές που θα μπορούσαν να έχουν μια επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή του εμπορίου, της ανάπτυξης υπαίθρου κλπ. Είναι αλληλοσυμπληρωματικές υπέρ των φτωχών χωρών και βοηθούν να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των πολιτικών πέρα από τους αναπτυξιακούς στόχους. Η πολιτική της μετανάστευσης η οποία μας συνενώνει εδώ προφανώς είναι μείζονος σημασίας γιατί ασχολείται με σχέσεις μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών. Σε εποχές κρίσης όπως είναι αυτή η εποχή όπου αντιμετωπίζουμε η οικονομική, μια οικονομική κρίση ε, στρεφόμαστε προς τα έσω ενώ θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί και να έχουμε μια παγκόσμια προσέγγιση. Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, θα συνεχίσει και θα πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίε που μας παρέχει όσον αφορά τις πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσει και ευεργετήματα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακοί αριθμοί και οι στατιστικές που είδα τις προάλλες. Μόνο 5% του ποσού των πακέτων σωτηρίας των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα θα αρκούσαν για να πληρώ, να ε, χρηματοδοτήσουμε την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής χιλιετίας. Άρα υπάρχουν τα χρήματα. Η μετανάστευση είναι ένας τομέας πολιτικής, αλλά ε, παρέχει και θετικά υποδείγματα για την συνεισφορά για τη μείωση της φτώχειας στον πλανήτη. Όταν τα μεταστατικά ρεύματα γίνονται αντικείμενα σωστής διαχείρισης, τόσο οι πλούσιες χώρες, οι χώρες προ... προορισμού και οι χώρες προέλευσης μπορούν να υποφεληθούν. Ε, και μπορεί να συνεπάγεται μεγάλη βοήθεια στις ε, χώρες όπου χρειάζονται άτομα με υψηλές δεξιότητες. τα εμβάσματα από τους μετανάστες είναι μια άλλη θετική συμβολή. Αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα ε, ανέρχονται, ισοδυναμούν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανά έτος ε, που αντιστοιχούν σε αυτά τα εμβάσματα και μπορούν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των εξωτερικών σοκ και της κρίσης στον πληθυσμό. Και πολλά από αυτά τα κονδύλια θα μπορούσαν να επενδυθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει το κόστος αυτών των ε, συναλλαγών τους ώστε να γίνουν ταχύτερες και πιο ασφαλείς. Το Αφρικανικό Ινστιτούτο Εμβασμάτων εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και βρίσκεται υπό την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης και ε, δουλεύει σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και πραγματικά θα εξυπηρετήσει αυτή την καλύτερη ροή των βασμάτων προς την Αφρική. Αυτές οι οικονομικές ροές ευεργετούν πολλές οικογένειες ε, που βρίσκονται πίσω στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και η επίπτωση στην ευημερία τους είναι άμεση. Αλλά όλο και περισσότερο γυναίκες ε, μεταναστεύουν επίσης και όταν το κάνουν φαίνεται ότι το δικό τους επίπεδο βασμάτων είναι υψηλότερο και το αποστέλουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη μα στη χάραξη των πολιτικών μας. Πέρα από τη σημασία αυτών των οικονομικών συναλλαγών ή μεταφορών εμβασμάτων μάλλον που είναι ιδιωτική φύσεω, θα ήθελα να μείνω στη συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών προορισμού μέσω δικτύωσης, ε, μέσω ε, ε, επένδυσης σε προγράμματα ανάπτυξης. Ε, υπάρχουν σημαντικοί φορείς ανάπτυξης και τα 17 εκατομμύρια ευρώ ε, τα οποία επενδύθηκαν από την Επιτροπή θα ε, συνεισφέρουν στην υποστήριξη των χωρών προέλευση. Μία από τις προτεραιότητες μας συγγνώμη, είναι να έχουμε ένα διαφορεμένο διάλογο με αυτούς τους φορείς. Οι χώρες προορισμού επιτρέπουν έχουν τη δυνατότητα μέσω των μεταναστών να αναπτύξουν πολλούς τομείς της οικονομίας τους. Και αυτό είναι ένα τομέα που θα πρέπει να ε, φωτίσουμε για την κοινή γνώμη σε εποχές κρίσης. Γιατί πράγματι οι οικονομικοί τομεί, όπω είναι η δημόσια υγεία, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες λοιπά ε, δείχνουν τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις δικές μας χώρες. Και αν λάβουμε υπόψη αυτές τις πολλαπλές επιπτώσεις ε, στον ορισμό των δημόσιων πολιτικών σε σχέση με τη μετανάστευση προϋποθέτει μια αναθόρηση της διαδικασίας χάραξης πολιτικών που πολύ συχνά είναι περιοριστικές και περιορίζονται στην πολιτική δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. Σήμερα η πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, ανάπτυξης, απασχόλησης και επίσης οι Υπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διατύπωση αυτών των πολιτικών και στη χάραξη αυτών των πολιτικών. Και αυτό που κάνουμε σήμερα με αυτή την κοινή συνδιάσκεψη των χωρών ΑΚΕ, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου, που όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την ε, χάραξη αυτής της πολιτικής με μεγαλύτερη ελεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ε, οργανώσεων και θεσμικών οργάνων που τελικά συμμερίζονται τους ίδιους στόχους. Μια συνεκτική πολιτική θα δώσει μια όθηση σε μια σφαιρική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση. Σκοπό που υιοθετήθηκε το 2005 και στοχεύει στην ε, συνεργασία με τις τρίτες χώρες όσον αφορά θέματα όπως είναι η χορήγηση ασύλου κλπ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πίσω ότι η Αφρική και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν μια στρατηγική εταιρική σχέση από το 2007 στη Λισαβόνα που μας δίνει τη δυνατότητα στη βάση ενός εντατικοποιημένου διαλόγου να ανταπεξέλθουμε στις κοινέ προκλήσεις. Η εταιρική σχέση έχει τη δυνατότητα να, ενισχύσει και να προωθήσει τη συνεκτικότητα των πολιτικών και μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετανάστευση και απασχόλησης εμπορίου Ειρηνή, ασφάλεια και ανθρώπινων δικαιωμάτων, θέματα τα οποία ε, παραδοσιακά ήταν μεμονωμένα. Και αυτό εντό του μοναδικού πλαισίου συνεργασία στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη και στην Αφρική. Ε, το brain drain, η φυγή των εγκεφάλων, ε, φαινόμενο που παρουσίασε ο κ. Πέτερν, είναι ένα άλλο πολιτικό και ιδιαίτερο σε βάση στο θέμα. Η Κομισιόν έκανε μια σειρά προτάσεων, ιδιαίτερω για να υποστηρίξει τον ορισμό των πολιτικών που ευεργετούν την ε, παραμονή εξειδικευμένου προσωπικού στις χώρες προέλευσης που είναι πολύ σημαντικό. Οι πολιτικέ αυτέ βασίζονται στην κατάρτιση, στην παροχή κινήτρων, καθώ και στι πολιτικέ ε, πρόσληψεις. Αυτέ οι προσεγγίσει είναι ιδιαίτερα σημαντικέ για την Αφρική, γιατί δίνουν στην Ήπειρο αυτή με τεράστιο ε, δυναμικό και ανθρώπινου πόρου, παρά την ανάγκη υψηλή κατάρτιση να διατηρήσει το δυναμικό της ε, και ε, υποβοηθούν τον έλεγχο αυτού του φαινομένου της φυγής εγκεφάλων. Η δημιουργία Ινστιτούτων ε, Διαχείρισης σε χώρες όπως είναι το Μαλί είναι μία από τις απαντήσεις που προτείνουμε από τη δική μας πλευρά και θα μπορούσαμε αργότερα να συζητήσουμε ε, με τους εταίρους μας από το Μαλί που είναι παρόντες εδώ σήμερα. Αυτή είναι μόνο η επαρχή και αυτός ο τύπος πρωτοβουλειών θα στεφθεί από επιτυχία εφόσον μπορούμε να αυξήσουμε τη νόμιμη μετανάστευση και τις δυνατότητες νόμιμης κινητικότητας. Είναι σημαντικό αυτή η πτυχή μιας σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης να εφαρμόζεται ε, ακριβώς όπως άλλες ε, πτυχές ε, πρόχειται του ιδίου, της ίδιας προβληματικής. Η συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη είναι ιδιαίτερος σημαντικός παράγων, ούτως ώστε να μπορούμε να δρούμε με έναν συνεκτικό τρόπο για να ανταποκρινόμαστε στις παγκόσμιες θα πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια για μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Και βεβαίω αυτό δεν είναι εύκολο έργο και είναι αναγκαία αυτή η παραπάνω προσπάθεια ε, και η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων της χιλετίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you, uh, Vice President Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο κύριε Βάλστρομ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή του πρώτου πάνελ, τον βοηθό Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Μάριο Αμάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πέτερη, κυρία Βάλστρομ, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Πρόεδρο Πέτεριν και την ε, Επίτροπο Βάλστρομ που τόνισαν τη σημασία του ρόλου των, ε, ε, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, των βουλευτών, όταν συζητάμε και προωθούμε την συνοχή στις πολιτικές ανάπτυξης. Το θέμα της συνοχής της πολιτικής ανάπτυξης και της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτού του δύσκολου καιρού, καθώ και οι αναπτυσσόμενε και οι αναπτυγμένες χώρε ε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν οικονομική και οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τη γοργή άνοδο της, απα... της ανεργίας. Η συνοχή για την αναπτυξιακή πολιτική είναι δύσκολη ακόμα και στις παχές αγελάδες. Επομένως, χρειάζεται να κάνουμε διπλές προσπάθειες για να την εξασφαλίσουμε στις συχνές αγελάδες. Ο, ο κάνει ό,τι μπορεί για να συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια ανταπόκρισης και καταπολέμησης της κρίσης. Δημοσιεύσαμε πρόσφατα την στρατηγική μας απάντηση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τονίσαμε τις προσπάθειες ε, που κάνουμε για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση και να αδράξουμε την ευκαιρία για να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή καθαρή και δίκαια παγκόσμια οικονομία. Οι επιπτώσει τη κρίση στι αναπτυσσόμενε χώρε θα επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη των χωρών του ΩΣΑ και η πρόοδο για τη μείωση τη στόχιας μπορεί να ακυρωθεί. Ο Γενικό Γραμματέας μα, ο κ. Γκούρια, λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να παραστεί σε αυτή τη διάσκεψη και ο πρόεδρο ε, τη Επιτροπή ΔΑΚ, ο κ. Ντόιτσερ, θα σα μιλήσει σε λίγο και ζήτησε τον περασμένο Οκτώβριο από του βασικού δωρητέ να τιμήσουν τις αναπτυξιακές τους δεσμεύσεις παρά την οικονομική ύφεση. Οι κυβερνήσεις που ανήκουν στην Επιτροπή DAX συμφώνησαν να διατηρήσουν τις αναπτυξιακές ροές με βάση τις δεσμεύσεις τους. Το να αποφύγουμε τον προστατευτισμό και το να κρατήσουμε ανοιχτό το παγκόσμιο εμπόριο είναι άλλα βασικά στοιχεία για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ σημαντικό τμήμα της ανάπτυξης αλλά δυστυχώς είναι μόνο ένα τμήμα αυτής της εικόνας. Γιατί είναι σημαντική η συνοχή της αντιξιακής πολιτικής. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ως προς το τι σημαίνει η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και γιατί πιστεύουμε ότι είναι όλο και πιο σημαντικό θέμα για τους πολιτικούς. Σε μια ελεοξαρτώμενη παγκόσμια οικονομία, οι επιπτώσεις των πολιτικών που θέτουν και εφαρμόζουν οι χώρες του ΟΣΕ, του ΟΣΑ συγγνώμη, και οι αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία ε, θα έχουν ε, παγκόσμια εμβέλεια. Επομένως, για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μείωσης της παγκόσμιας στόχιας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τους για θέματα τα οποία ξεπερνούν τη βοήθεια, υποστηρίζουν ή τουλάχιστον δεν υποσκάπτουν τις αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτό σημαίνει η συνοχή της ε, αναπτυξιακής πολιτικής. Εσείς ως πολιτικοί ξέρετε πολύ καλά ότι στις εθνικές συζητήσεις οι ανησυχίες όπως η ενδυνάμωση της ασφάλειας ή η τόνωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας ε, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τη μείωση της στόχιας. Για τους πολιτικούς που προσπαθούν να εξορροπήσουν τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων συμφερόντων, η ανάγκη συνοχής της πολιτικής ανάπτυξης μπορεί να μην είναι τόσο προφανής. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι πλήρης συνεπείς πολιτικές μπορεί να μην είναι εύκολο πολιτικά ή εφικτό πολιτικά, αλλά οι μη συνεπείς πολιτικές είναι αναποτελεσματικές όποιος στόχος και αν είναι πρώτος στην ατζέντα μας και η έλλειψη συνοχής ε, κοστίζει στους ε, φορολογούμενους και στους στοχούς των αναπτυσσομένων χωρών. Επιπλέον, το να παραμελήσουμε την αναπτυξιακή διάσταση είναι κοντόθωρο και μακροπρόθεσμα θα υποσκάψει την υλοποίηση άλλων στόχων όπως τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια ή τους περιβαλλοντικούς στόχους. Όπως λέει η έκθεση του ΟΣΑ για την αναπτυξιακή συνεργασία το 2007, όλες οι χώρες παραθέτω, έχουν ένα κοινό συμφέρον για να επιτύχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες βιώσιμη και ευρεία ανάπτυξη. Οι πολιτικές οι οποίες υποσκάπτουν τους αναπτυξιακούς στόχους ε, είναι επί παραδείγματι οι γεωργικές επιδοτήσεις, οι κλιματικές αλλαγές, η υπερβολική εκμετάλλευση των λευτικών πόρων, η μετανάστευση των ε, επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η διατήρηση ε, εμπορικών περιορισμών. Ο ΩΣΑ έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της συνοχής της αντιξιακής πολιτικής ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1990. Ο ΩΣΑ έχει εξηγήσει τη σημαντική συσβολή, συνεισφορά που μπορεί να έχει αυτή η συνοχή στο να ενδυναμώσει την ε, ανάπτυξη και να μας δώσει διάφορα στοιχεία για την αναπτυξιακή διάσταση στο εμπόριο, στη γεωργία και στη μετανάστευση κτλ. Το να μαθαίνουμε από του ομοίου μα και να πιεζόμαστε από του ομοίου μα ε, ήταν αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόθεση τη ε, συνοχή τη αντιξιακή πολιτική. Πέρυσι τον Ιούνιο οι Υπουργοί του ΟΣΑ υιοθέτησαν την Υπουργική Δήλωση για την ε, συνοχή τη αναπτυξιακή πολιτική. Στην κοινοτική διόγλωση αυτό σημαίνει ότι η συνοχή τη αναπτυξιακή πολιτική είναι τώρα κεκτημένο του ΟΣΑ. Η δήλωση τονίζει το στοιχείο ότι η συνοχή της αναπτυξιακή πολιτικής είναι βασικό στοιχείο για να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις με βιώσιμο τρόπο. Οι Υπουργοί τόνωσαν εκ νέου την δέσμευσή τους στο να συνεχιστούν οι προσπάθειες ούτω ώστε οι αναπτυξιακοί στόχοι να ληφθούν υπόψη σε τομείς όπως η μετανάστευση. Τώρα, η μετανάστευση και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί η μετανάστευση είναι σημαντική για την συνοχή τη αναπτυξιακή πολιτική. Καταρχάς, γιατί οι ευρείε πολιτικές μπορεί να αυξήσουν τα ωφέλη της μετανάστευσης από την αναπτυξιακή πλευρά. Δεύτερον, γιατί η μετανάστευση δείχνει κάποιες από τις μεγάλες πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες που προσπαθούν να προοδεύσουν προς μια συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική αν διαχειριζόμαστε σωστά την ε, εργατική μετανάστευση, αυτό μπορεί να είναι υποφελέ για τι χώρε προορισμού και μπορεί να είναι και σημαντικό και για τι χώρε προέλευση. Τα εμβάσματα έχουν δείξει ότι βελτιώνουν πολύ σημαντικά την ευημερία αυτών που τα λαμβάνουν και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επενδύσει στην εκπαίδευση και στην υγεία. Η επιστροφή στη χώρα προέλευση μπορεί να συνδεθεί με μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας με επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και με την αγορά εργασίας στις χώρες προέλευσης. Είναι προφανές ότι το μέγεθος της συνεισφοράς ε, παίζει από χώρα σε χώρα. Είναι μεγαλύτερο στις μικρές χώρες όπου οι μετανάστες είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, όπως ε, παραδείγματος χάρη σε κάποιες ε, κεντροαμερικανικές χώρες, χώρες Καραϊβικής και του Ειρηνικού ειδικά νησιά του Ειρηνικού, όπου τα εμβάσματα είναι σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ. Σε άλλες χώρες οι επιπτώσεις είναι πιο τοπικές. Τα εμβάσματα είναι τμήμα των ιδιωτικών ροών και επομένω η χρήση τους εξαρτάται από τις ιδιωτικές αποφάσεις. Αλλά αυτές οι αποφάσεις εξαρτώνται με τη σειρά τους από εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να αυξήσει τις ε, ευκαιρίες απασχόλησης στις αντισόμενες οικονομίες, αλλά μπορεί να μην μειώσει τη μετανάστευση βραχυπρόθεσμα, καθώς περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να μετακινηθούν, να φύγουν. Επομένως, ε, μπορεί η οικονομική επιτυχία μπορεί να συνοδευτεί από περισσότερους διεθνείς μετανάστες. Κατά συνέπεια, η μετανάστευση είναι μία από τις πολλές παραμέτρους και τα κανάλια μέσα από τα οποία οι πολιτικές των χωρών του ΩΣΑ μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια, οι πολιτικές μετανάστευσης είναι σημαντικές στις συζητήσεις για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Μετανάστευση, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Τρία σημαντικά αποτελέσματα που συνδέονται με την οικονομική κρίση μπορούν να αναφερθούν. Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας πρώτον, τα εμβάσματα και οι καθαρές μεταναστευτικές ροές. Από την ε, παρελθούσα εμπειρία προκύπτει ότι οι μετανάστες είναι οι πιο ε, έντονα πληττόμενοι στην αγορά εργασίας όταν υπάρχει ύφεση. Ε, χάνουν πρώτοι τις δουλειές τους. Οι μετανάστες επίσης έχουν, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τους ημεδαπούς που αναζητούν απασχόληση ή που και βρίσκουν τις χειρότερες δουλειές όταν περάσει η ύφεση. Η υπερβολική ανάπτυξη των εμβασμάτων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει ή έχει αντιστραφεί σε ορισμένε χώρε. ταυτόχρονα, η, τα εμβάσματα και οι ροέ από τα εμβάσματα είναι λιγότερο ασταθεί από ότι τα εισοδήματα από τις εξαγωγές ή από τις ε, κεφαλιακές ροές, τα οποία έχουν ε, καταρακωθεί. Παρ' όλα αυτά, τα εμβάσματα ε, θα δυσκολέψουν ε, λιγότερα εμβάσματα θα δυσκολέψουν τα πράγματα για τις οικογένειες και τις ε, κοινότητες στις πατρίδες των μεταναστών. Θα πάνε οι μετανάστες όμως σπίτι. Οι χειρότερες αναπτυξιακές προοπτικές στις χώρες και προοπτικές απασχόλησης στις χώρες ΟΣΑ μπορεί να μας οδηγήσουν στο να πιστέψουμε ότι θα οδηγήσει αυτό τους μετανάστες πίσω στις πατρίδες τους. Αλλά από τα στοιχεία που έχουμε ε, δεν ξέρουμε ε, εάν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Η οικονομική κρίση έχει καταστήσει την ε, εργατική μετανάστευση μια χαμηλή προτεραιότητα στις χώρες όσα. Όμως η γύραση θα παραμείνει μαζί μας και οι εργατικές ανάγκες θα επανέλθουν όταν επανέλθει και όταν εξαλειφθεί μάλλον η ύφεση. Οι χώρες του ΩΣΑ πρέπει να μην ξεχνάνε ότι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ε, τις δημογραφικές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαζόμενο να, να παρατείνουν την, ε, το χρόνο σύνταξης, να αντιστρέψουν την ε, εκρηκτική ανάπτυξη των ε, ανθρώπων που είναι άρρωστοι και ανάπηροι και να βελτιώσουν και να αυξήσουν την εκπαίδευση των ενηλίκων, την διαβίου μάθηση και να αυξήσουν την παραγωγικότητα με κάθε δυνατό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βασιστούν και στους μετανάστες. Είναι αναπόφευκτο λοιπόν προκειμένου να έχουμε μία... Να τους έχουμε υπόψη, να θέλουμε να έχουμε ε, λειτουργικές πολιτικές. Η κρίση λοιπόν μόνο ε, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα. Ε, τώρα, οι δημόσιες συζητήσεις για την μετανάστευση από τους πολιτικούς και από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων πρέπει να είναι παραδειγματικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λέμε και τα κακά νέα, αλλά θα πρέπει να λέμε στον πληθυσμό μας, στους πολίτες μας, ε, σωστά πράγματα, να τους περνάμε τα σωστά μηνύματα για τη θετική συνεισφορά των μεταναστών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Είναι πολύ εύκολο κάποιοι να κατηγορούν τους μετανάστες ε, για να κερδίσουν ε, την εύνοια του κόσμου. Αλλά είναι ο ρόλος των βουλευτών και των οργανώσεων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΑ να βλέπουν προς τα εμπρός, προς το μέλλον. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καλύτερες αποφάσεις ε, δεν λαμβάνονται εν το μέσο μιας κρίσης, παρότι πρέπει να ληφθούν. Η δουλειά μας είναι να σκεφτούμε παραπέρα, μακροπρόθεσμα, η επίπτωση της κρίσης στη μετανάστευση και τα μέτρα υποεξέταση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό τομέα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, καθώς οι κοινωνικές αναταραχές ε, γίνονται όλο και πιο αισθητέ. Συζητήσει όπως αυτές που έχουμε σήμερα μεταξύ πολιτικών από διάφορες χώρες και υπήρους είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να δημιουργήσουμε ευρύτερε συμμαχίες και να μάθουμε η μένα τους δε. Επίσης ε, τονίζουν την, ε, το, το, θέμα της μετανάστευσης που είναι παγκόσμιο και που απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα ακόμα βήμα στην παραδοσιακή συνεργασία ΩΣΑ Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε αυτέ προκλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αμάνο. Θα δώσω το λόγο σε δύο ακόμη προσκεκλημένους ομιλητές θα ήθελα όμως να του ζητήσω αν είναι δυνατόν να μειώσει το χρόνο ομιλίας τους κατα δυο δύο-τρία λεπτά ο καθένας τους ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε στις 12.30. Εντάξει, μπορούμε να μείνουμε λεπτά λεπτάκια ακόμη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Εκχατόιτσερ ε, πρόεδρος της ε, περίφημης επιτροπής DAC του ΩΣΑ ε, της ε, βοήθειας στην ανάπτυξη επιτροπής βοήθειας στην ανάπτυξη δηλαδή ήταν επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος του Ινστιτούτου στην Κωνσταντίνα για τη Δημοκρατία στη Λατινική Αμερική. Κύριε Ντόιτσερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι χαίρομαι ιδιαίτερα από το θέμα της συνεκτικότητας των πολιτικών ε, αποκτά όλο και περισσότερη σημασία πιστε, είμαι πεπισμένος για την σημασία της ανάγκη να υπάρχει αυτή η συνεκτικότητα για τις πολιτικές της ανάπτυξης φαντάζομαι και της μετανάστευσης αλλά έχω και άλλη μια βαθιά πεποίθηση ε, τα τελευταία και είναι, η οποία είναι η εξή ότι ο τομέας της ανάπτυξης και της βοήθειας στην ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια δεν συνεργάστηκε όσο έπρεπε με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή ε, συνάντησή μας εδώ. Έχω ακόμη 12 λεπτά μου λένε. Θα προσπαθήσω λοιπόν σε αυτά τα 12 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να σας πω, να κάνω μερικά σχόλια για το θέμα που σας απασχολεί σε σχέση όμως με την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουν ε, να ασχοληθούν οι δωρητές. Ε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται. Πριν από μερικούς μήνες υπήρχε η άποψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα επηρεαστούν από την χρηματοπιστωτική κρίση που θα πλήξει τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν και σήμερα πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντικός κίνδυνος οι αναπτυσσόμενες χώρες να είναι τα χειρότερα θύματα της κρίσης αυτής. Τι ποιας κλίμακας κρίση μιλάμε με, ό, όταν ε, ξέρουμε από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι μείωση στην ανάπτυξη κατά 1% σημαίνει 20 ακόμη εκατομμύρια άτομα που μπαίνουν, ζουν σε συνθήκες φτώχειας θα πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή η ανάπτυξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 3,7 του 2007 έπεσε στο 0,5 όπως προβλέπετε το 2009 70 ε, ακόμη ακόμη άτομα θα ζουν στις συνθήκες φτώχειας πέρα των 100 που ήδη βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Όλες οι πρόοδοι που έγιναν τα τελευταία χρόνια λοιπόν θα καταρρεύσουν, θα αντιστραφούν δυστυχώς και τα πράγματα ε, συνεχώς ε, φαίνεται να δυσκολεύουν και οι κασάνδρες ανά τον κόσμο προβλέπουν όλο και περισσότερο και χειρότερη, χειρότερες εξελίξεις. Είναι λοιπόν πολύ, μεγά, πολύ κρίμα που θα χάσουμε ό,τι κερδίσαμε στον τομέα της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Και τώρα θα ήθελα με δύο λόγια να μιλήσω για τα το πώς δρά ο ΣΑ ε, και πώς ε, και από οικονομική άποψη ε, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι πάρα πολλές εκτός από την βοήθεια η οποία δίνεται πάρα πολλά άλλα οικονομικά μέσα εξαγωγές, ε, βάσματα κτλ θα πληγούν για αρχίζω με τις εξαγωγές σε σχέση με, τις, με τα παλιά χρόνια βλέπουμε μια πραγματική ανατροπή των τάσεων πρώτη φορά γίνεται αυτό μετά την ε, ε ύφεση του 1982 άρα ε, τα πράγματα δεν είναι καλά από εκεί και πέρα για τις οικονομικές ροές του ιδιωτικού τομέα ε, από ένα δολάρια το 2007 το 2008 βρισκόμαστε μονάχα στα 500 δις και έκτοτε το 2009 βλέπουμε μια περαιτέρω πρωτόση στα 165 δις δολάρια δηλαδή μείωση πάνω από 80% σε σχέση με το 2007 για κάποιες χώρες χαμηλού εισοδήμα χαμηλών φτωχές όπως παραδείγματος χάρη είναι η Κένια ή η Γκάνα αυτό είναι τραγικό η ε, οι χώρες αυτές λειτουργούσαν καλά, είχαν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με τις κεφαλαγορές της διεθνής. Αυτή τη στιγμή χάνουν τα κέρδη αυτά που είχαν. Τώρα έρχομαι στα εμβάσματα, τα οποία επίσης θα υποφέρουν, δεδομένου ότι τα έσοδα των μεταναστών θα πέσουν εφόσον θα αυξηθεί η ανεργία. Και ιδιαίτερα στις για τις φτωχές χώρες όπου τα εμβάσματα είναι ένα μεγάλο μερίδιο των ε, κρατικών εσόδων τα πράγματα θα είναι προφανώς χειρότερα και τώρα έρχομαι στη βοήθεια γιατί προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να και η έννοια της βοήθειας να Επιπρέαστη αρνητικά από την κρίση. Μετά την ύφεση του 1991-1992 η ε, επίσημη βοήθεια που δινόταν ε, έπεσε κατά 22% και μέχρι το 2003 Μόνο το 2003 μπόρεσε να ξανανεύει στα προηγούμενα επίπεδα. Αλλά η σημασία της βοήθειας αυτής νομίζω ότι εντείνεται, επιτείνεται από την χρηματοπιστωτική κρίση που διανύουμε. Γιατί ε, δεδομένου ότι άλλες πηγές χρηματοδότησης θα περικοπούν, θα ε, ε, μειωθούν το μόνο που απομένει είναι η βοήθεια για, κάθε, για κάποιες χώρες ή για τις φτωχές χώρες είναι το, η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης το 2005 και 2006 η βοήθεια αυτή ήταν 48 δις δολάρια που ήταν διπλή τεράστιο διπλάσιο ποσό από ότι τα έσοδα από το εμπόριο και τα εμβάσματα μαζί παραδείγματος χάρη. Όπως είπε ήδη ο κύριος Αμάνο, ε, επαναλαμβάνω και εγώ ότι ζητούμε από τις χώρες της, Επιτρο... της Επιτροπής ΝΤΑΚ και από όλες τις χώρες να υποσχεθούν βοήθεια, να δώσουν μια επίσημη υπόσχεση βοήθειας. Ο ναι, και να συνεχίσουν να σέβονται τις υποσχέσεις που έδωσαν στο παρελθόν δεν είναι σωστό να γίνει αυτό που έγινε σε προηγούμενες περιόδους ύφεση, όπου μειώνονταν ο προϋπολογισμός τα κονδύλια για τη βοήθεια έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις πρέπει να αντιστηρίσουμε και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι φτωχές χώρες συνεχίζουν να εξαρτώνται από την εξωτερική στήριξη και η εξάρτηση αυτή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι άλλες πηγές χρηματοδότηση όπως είπα πέφτουν. Οποιαδήποτε μείωση θα ήταν τραγική. Και θα κάνουν ακόμη πιο ευάλωτες κάποιες χώρες που είναι ήδη φτωχές και ευάλωτες. Αν κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω, το 2008 πραγματικά ήταν ένα έτος κρίσεων. Η κρίση στα τρόφιμα, η κρίση στα καύσιμα και τώρα η χρηματοπιστωτική κρίση. Όλες αυτές είναι παγκόσμιες κρίσεις. Όλες άρα απαιτούν παγκόσμιες διεθνείς λύσεις και έδειξαν ο, οι κρίσεις όλες αυτές ότι οι μεμονωμένες αντιδράσεις ή λύσεις όπως νομίζουν ορισμένοι δεν βοηθούν. Χρειάζονται λοιπόν παγκόσμιες λύσεις οι στις οποίες να συμμετέχουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες μπορούν να ξέρουν πώς αυτές οι λύσεις θα εφαρμοστούν στο εσωτερικό τους. Οι εθνικές πολιτικές συνεχίζουν να υστερούν σε σχέση με την πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο αν θέλουμε να δουλέψει η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να λειτουργήσουν τα πολυμερή συστήματα συνεργασίας. Οι κρίσεις που ζήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά και είναι τεράστια σημασία αν αυτό που λέω αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα στον πλανήτη γι' αυτό και για τούτη εδώ τη χρηματοπιστωτική κρίση η συνεργασία ε, στην ανάπτυξη πρέπει να είναι σημείο κλειδί που δεν είναι λόγο κάποιος μόνος του μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα η πολιτική η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ να ανοί, γίνει πιο ανοιχτή στην πραγματικότητα των παγκόσμιων αλλαγών και προκλήσεων γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο και θέλω να το τονίσω αυτό η συνεκτικότητα των πολιτικών και οι προσεγγίσεις, οι φιλοσοφίες που θέτουν οι διάφορες χώρες στις οποίες να συμμετέχει ολόκληρη η κυβέρνηση. Η πριν από μερικές εβδομάδε η Επιτροπή μας ΝΤΑΚΑ αποφάσισε να κοιτάξει δύο, τρία συγκεκριμένα θέματα με σε περισσότερο βάθος στο το εμπόριο, το περιβάλλον και τη μετανάστευση. Και κλείνοντας τώρα θα ήθελα όπως είπε και ο Πρόεδρος να συμφωνήσω απόλυτα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπενθυμίσω και εγώ τις κυβερνήσεις των χωρών δωρητών ότι έχουν αναλάβει υποχρεώσεις. Χρειαζόμαστε παγκόσμια συνεργασία, χρειαζόμαστε ε, συνεκτικές πολιτικές και χρειαζόμαστε επενδύσεις στην συνεργασία, στην ανάπτυξη για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Now the floor Τώρα το λόγο έχει ο κύριος David Arkless που είναι πρόεδρος του Global Corporate Affairs έχει μία ιδιαίτερως μακρά εμπειρία στον τομέα της ε, βοήθειας προς τις χώρες για να αναπτύξουν τις ε, ε, στρατηγικές της αγοράς. Υπήρξε σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων και τώρα είναι μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού για, για τη Μετανάστευση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είναι καλό που βρίσκομαι εδώ σήμερα το πρωί. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, διακεκριμένα μέλη. Ε, δεν ξέρω και αν υπάρχουν κάποιοι μη ειδικοί, θα ήθελα να τους κολοημερίσω και αυτούς. Ε, το ανθρώπινο δυναμικό είναι ε, οι εργοδο... Ε, έχουμε 5 εκατομμύρια εργοδοτών και αντιπροσωπεύει μία ε, συνιστόσα. Εκπροσωπώ τη Manpower. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος εργοδότης και βεβαίως ε, η εργοδοσία είναι πολύ ε, σημαντική αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης. συμμετείχα στο φόρουμ του Νταβός και ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο. Ε, Χθε μόνο ήμουν στο Μεξικό και θα μπορούσα να σας πω ε, ποιες είναι οι επιπτώσει αυτής της κρίσης για τους συνηθισμένου ανθρώπους και ποιε είναι οι επιπτώσει στην μετανάστευση. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν 250 εκατομμύρια μετανάστες σε ολόκληρο του κόσμου και ο αριθμός θα αυξηθεί σε 400 εκατομμύρια. Οι λόγοι μετανάστευση είναι προφανής, η κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές και κατά δεύτερο λόγο ε, οι πολιτικές σειράξεις, οι πολιτικές συγκρούσεις και τέλος οικονομικοί λόγοι. Και αυτό δεν θα πάυσει γιατί τα οικονομικά επίπεδα θα διαφέρουν στα διάφορα μέρη του κόσμου. Για ανθρώπους που κινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο για να εργαστούν υπάρχουν επίσημα, επίσημα και μη επίσημα εμπόδια. Και θα ήθελα να σας τα περιγράψω. Η μετανάστευση για την εργασία συνήθως θεωρείται θετικό ε, σε περιοχές ανάκαμψης αλλά αρνητικό σε εποχές κρίσης πώς σχετίζεται με την ανεργία, γιατί το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στα γραφεία μας, στα 5.000 γραφεία μας. Οι πρώτοι άνθρωποι που πετιούνται έξω από τη δουλειά τους είναι αυτοί που αμείβονται χαμηλά και δεν έχουν πολλά προσάντα. Τι συμβαίνει στους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί γίνονται μακροπρόθεσμα άνεργοι. Για ποιο λόγο γιατί δεν κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους εργαζόμενους μετανάστες. Τελικά έχουν δύο επιλογές, χάνουν τη δουλειά τους και είτε μπορούν να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται είτε μπορούν να φύγουν. Και το να φύγουν σημαίνει να πάνε σε μια άλλη χώρα όπου μπορούν να εργαστούν ή μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους. Συχνά υπάρχουν επίσημα ή ανεπίσημα εμπόδια για αυτές τις επιλογές και συνεπώς υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Να μην ξεχνάτε ότι δεν μιλούμε μόνο για διασυνοριακή μετακίνηση εργαζόμενων εδώ, αλλά υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια εκατομμύρια εσωτερικών εργαζόμενων που μετακινούνται σε χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία. Και αυτός ο αριθμός ε, και ο αριθμός αυτός των ε, μεταναστών θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Ε, θεωρούμε ότι η αύξηση έχει τρομακτικές επιπτώσεις σε μια νέα κατηγορία ανθρώπων που τους ε, ονομάζουμε αστικούς μετανάστες, αστικούς πρόσφυγες. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα 13 εκατομμύρια Κινέζων την πρωτοχρονιά έχασαν την ε, δουλειά τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Στην Ισπανία υπάρχει αύξηση 70% της ανεργίας και η κυβέρνηση δίνει κίνητρα, οικονομικά κίνητρα επιστρέψει στις πατρίδες τους, αλλά ε, αρνούνται να το κάνουν. Στην ε, Νορβηγία πληρώνουν τα εισιτήρια των λεωφορείων για ανθρώπους από την Ανατολική Ευρώπη για να επιστρέψουν στις χώρες τους και αρνούνται αυτοί να το κάνουν. Επίσης στο Μεξικό Σημαίνουν ε, Συμβαίνουν ανάλογα φαινόμενα. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνει dumping σε 250.000 ε, ανθρώπων που βρίσκονται στο Χουαρέζ προκειμένου να επιστρέψουν στην, Ισπα... πατρίδα του στο Μεξικό. Αλλά αυτοί αρνούνται να το κάνουν γιατί πολλές φορές δεν μιλούν καν Ισπανικά ε, μας δίνουν όλα αυτά τις διαστάσεις του προβλήματος και ο αντέκτυπος είναι προφανής. Ε, οι χώρες προορισμού έχουν ένα τεράστιο φορτίο ε, και υπάρχει το λεγόμενο το φαινόμενο ξενοφοβίας έναντι ε, των εργαζόμενων. Τα ποστά των εμβασμάτων 27 εκατομμύρια από 18 στην Κίνα. Ε, ε, αυτή η μείωση είναι, η ισχύ των εμβασμάτων είναι τεράστια σε όλες τις χώρες. Φανταστείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις χώρες προορισμού. Ή στη Γαλλία για παράδειγμα από 12 δις τον περασμένο χρόνο σε 6 δις αυτό το χρόνο όσοι επαναπατρίζονται πολύ συχνά είναι ανεπιθύμητοι και προκαλούν φαινόμενα κοινωνικής αναταραχής και είναι τεράστιο φορτίο για χώρες όπου η ανεργία πολύ συχνά είναι πάνω από 13%. Ωραία, τι πιστεύουμε εμείς. Είμαστε εντελώς εξαρτημένοι με την κατάσταση αυτή. Γιατί, γιατί ακόμα να γίνεται λόγος για στόχους, ε, συνεκτική πολιτική, προδιαγραφές και ρυθμίσεις. Αλλά δεν υπάρχουν ε, ρυθμίσεις

πέρα από τις εθνικές χώρες που είναι υπεύθυνε για τη μετανάστευση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο διεθνή ευελιξία στον αφορά τους εργαζόμενους και αυτό σημαίνει παραγωγικότητα, σημαίνει μεγαλύτερο output, σημαίνει αύξηση της οικονομίας, σημαίνει μεγαλύτερο κύκλο κατανάλωσης κλπ. ώστε να είναι όλοι ευτυχείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κίνηση των εργαζόμενων και της εργασίας, η μετακίνηση είναι καλό πράγμα. Η εργασία είναι καλό όταν μετακινείται γιατί βοηθάει τις χώρες να αναπτύσσονται. Οι εργαζόμενοι είναι καλό όταν μετακινούνται γιατί μπορούν να έχουν μια αντιστάθμιση για τις καταστροφικές δημογραφικές τάσεις. Ε, η Ευρώπη χάνει τεράστιο ποσοστό των εργαζόμενων, 50 εκατομμύρια εργαζόμενους. Πού θα τους βρούμε το χρόνο. Ε, είναι καλό να στραφούμε σε τις χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή η Τουρκία, γιατί εκείνοι αυξάνουν τον πληθυσμό τους κατά 50 εκατομμύρια εργαζόμενους. Λοιπόν, υπάρχει έλλειψη ικανοποίηση ε, στις κυβερνήσεις. Οι μετανάστες αυξάνονται, μάλλον θα είναι 50 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Η, διακίνηση, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων 40.000 ε, παραπάνω άνθρωποι. Οι άνθρωποι γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση στην εργασία τους, συνεπή αυτών των φαινομένων. Τι κάνουμε λοιπόν. Προσπαθούμε εμείς να κινηθούμε μόνοι μας και να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις και τα, τους οργανισμούς. Το πρωτόκολλο της ε, Μανίλα ήταν θετικό σε σχέση με την διεθνή εργασία. Αλλά όταν προωθήθηκε στο Αμπουντάμπι πέρσι, τρεις Υπουργοί Εργασίας ε, και δύο στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, απολύθηκαν. Συνεπώς λοιπόν χρειάζεται πολύ τόλμη για να επιφέρει κανείς τέτοιες αλλαγές. Η, η πολιτική μετανάστευση χρειάζεται άμεση δράση. Ε, και θα υπάρχει και μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Στη, στο Βιετνάμ έχουμε μια κοινοπραξία με την κυβέρνηση για να βελτιώσουμε τα θέματα. Στην Κίνα παρέχουμε συμβουλές στην κυβέρνηση για τη χάραξη μιας λογικής πολιτικής εσωτερικής μετανάστευσης. Στην Αφρική προσπαθούμε να χειριστούμε τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα οι ε, οικονομικοί πρόσφυγες από τη Ζιμπάμπουε για παράδειγμα. Ε, προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πολλοί μας λένε ότι δεν είναι δική σας υπόθεση. Αλλά λυπούμεθα, είμαστε, είναι δική μας υπόθεση γιατί δεν υπάρχει το αρμόδιο πολιτικό πλαίσιο, το αντιδειγμένο πολιτικό πλαίσιο και εμείς τους αντικαθιστούμε. Εγώ δεν, είμαι, δεν, είμαι, δεν είμαστε πολύ δημοφιλείς λόγω των ξεκάθαρων απόψεων που έχουμε, αλλά πραγματικά δεν μας νοιάζει γιατί είναι δικές μας αυτές οι απόψεις και τις υπερασπιζόμαστε. Θα θέλαμε να κάνουμε το εξή, να αναγνωρίσουμε η αναγνώριση του δημοφραγραφικού προβλήματος τελικά ε, ε, δεν αρκεί. Ε, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Θα πρέπει να υπάρξει το πλαίσιο για την κυκλική μετανάστευση σε παγκόσμια κλίμακα. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι διμερείς συμφωνίες. Και παρακαλώ να δείτε να, σε αυτούς σαν ε, συνεκτικές ομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι χώρες του κόλπου. Την περασμένη εβδομάδα προσπάθησα να του πω θα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη συμφωνία εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει διμερείς συμφωνίε με την Ινδία, το Πακιστάν, την Κίνα, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες, το Μαρόκο και τον Μπαγκλαντές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ειδική συμφωνία με την Τουρκία και την Αίγυπτο. Γιατί την Αίγυπτο, γιατί έχει 93 εκατομμύρια ανθρώπων που πολλοί είναι άνεργοι. Θα του χρειαστείτε μελλοντικά στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος προς τα μπρό για μας μοιάζει ευθύς. Χρειάζομαστε πολλές διμερεί συμφωνίες, απουσία ενός παγκόσμιου πλαισίου. Και παρακαλώ να συμφωνήσετε τα εξή θέματα στο πλαίσιο αυτών των δημορών συμφωνιών. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, σωστά κριτήρια επιλογή και επιστοποίηση των ανθρώπων που κινούνται, προηγούμενη κατάρτιση των ανθρώπων πριν μεταβούν σε μια άλλη χώρα και πρωτόκολλο ανταλλαγή σε διαδικασίε ε, διέλευση των συνόρων. επίση προδιαγραφέ, ασφαλεία για του εργαζόμενου μετανάστε και κατάλληλοι μηχανισμοί επαναπατρισμού και επιστροφή, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους και να εισβάλλουν στην ανάπτυξη της δικής τους χώρας. Ε, δεν θα πρέπει η εξάπλωση εργασία να συνοδεύεται από κόστος, γιατί αυτό οδηγεί σε καταχρήσεις. Δεν θα πρέπει να γίνεται κατάσχεση των διαβατηρίων των ανθρώπων όταν πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα για να βρουν εργασία. Εμείς πιστεύουμε ότι από τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν. Υπάρχουν εν δυνάμει οι λύσεις και πραγματικά ο δρόμος, όπως σας είπα, είναι ευθύς, μια ευθεία. Uh, το γύρο του κόσμου. Ε? Πραγματικά, σας ευχαριστούμε για αυτό το πρόγραμμα εργασίας που μας προτείνετε. Και τώρα έχουμε χρόνο για τρεις παρεμβάσεις μόνο και τρεις απαντήσεις βέβαια. Μιλάμε για ανθρώπους ε, οι οποίοι έχουν ε, καταχωρηθεί, έχουν εγγραφεί έχουν πάρει αυτό το έντυπο, μπορούν να θέσουν ερωτήσεις λοιπόν και να πάρουν απάντηση. Οι... Όσοι δεν μπορέσουν να μιλήσουν το πρωί, θα μιλήσουν το απόγευμα. Όλοι όσοι έχουν εγγραφεί. Σήμερα το πρωί ε, έχουμε, θα ακούσουμε τρία άτομα. Τον Ιταλό γερουσιαστή καταρχήν. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άρκλες για την παρέμβασή του. Έθεσε πραγματικά τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργεί η μετανάστευση. Η λειτουργία της εταιρείας του ε, και ο ρόλος της ε, ε, ως ε, σύμβουλος διαφόρων ε, κυβερνήσεων θα έπρεπε να συμπληρωθεί από την προσπάθεια των ίδιων των κυβερνήσεων. Σήμερα δεν γίνεται καμία τέτοια προσπάθεια. Δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός όπου να εγγυάται τον τρόπο επιλογής, τις δεξιότητες των μεταναστών κτλ. Είναι μια τεράστια έλλειψη αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα των πολιτικών. Δύο προβλήματα που μου φαίνονται τεράστια, ανυπέρβλητα. Καταρχά η επίλυση του προβλήματος της λάθρομετανάστευση. Οι ΙΠΑ έχουν 12 έως 13 εκατομμύρια λαθρομετανάστες ε, στην επικράτειά τους. Ε, στην Ευρώπη με βάση εκτιμήσεις έχουμε 5-6 εκατομμύρια. Στην ε, Σοβιετική, πρώην Σοβιετική Ένωση 5 με 10 εκατομμύρια. Υπάρχει το εξή παράδοξο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει λαθρομετανάστες. Και σωστά. Αλλά δεν θέλει όμως και μαζικούς επαναπατρισμούς, μαζικές απελάσει. απελάσεις. Τι θα κάνουμε με αυτά τα 5, 6, 7 εκατομμύρια μεταναστών που έχουμε. Τι πολιτική συμβουλεύουμε στις κυβερνήσεις μας και στις χώρες μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Το πρόβλημα της κυκλικής μετανάστευσης. Υπάρχει μία τάση, σιωπηλή αλλά ισχυρή, να υποκαταστήσουμε την ε, μόνη μετανάστευση με την κυκλική μετανάστευση. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να δούμε την αρχική σελίδα της έκθεσης του ΟΣΑ του 2008 που μας λέει ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με αυτή την ε, κυκλική μετανάστευση. Δεν νομίζω ότι αυτή μπορεί να μας επιλύσει τα προβλήματα εργατικών ε, χεριών και εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή δυστυχώς calendario. Questo fa all'incirca il 20%. Νομίζω ότι είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δυστυχώς διακόπτουν τον ομιλητή. Η εκπρόσωπος από την Μπουρκίνα Φάσο. Euh, Καλημέρα σας από την Μπουρκίνα Φάσο. Εγώ είμαι το απτό παράδειγμα όλων αυτό που λέτε. Είμαι μετανάστρια που δούλεψε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Μπουρκίνα Φάσο για να δουλέψει σε μια άλλη εταιρεία ε, διεθνή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρος της Manpower. Για μας το βασικό πρόβλημα είναι πώς οι αποταμιεύσεις θα γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, πώς ε, η διασπορά θα ασχοληθεί με την χώρα προέλευσης. Διακόπτω το μικρόφωνο πάλι, συγγνώμη. Θα θέλαμε να, οι λύσεις να είναι γρήγορες, και ασφαλείς και παραγωγικές βέβαια. Θα θέλαμε επίσης να υπάρχουν κέντρα κατάρτισης, να δώσουμε έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς ε, στην επιχείρησή μου ε, προσπαθούμε να δώσουμε την έμφαση ε, στην κατάρτιση του πληθυσμού Έχουμε διάφορα εργαλεία. Ε, μας βοήθησε ο ιδιωτικό τομέας για να τα δημιουργήσουμε. Θα μας άρεσε να συνεργαστούμε με τη Manpower για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Δυτική Αφρική. Ένα κέντρο κατάρτισης ε, θα δημιουργηθεί στο Ουαγκαντούκου στην Ανατολική Αφρική. Ο Επίτροπος κ. Λουί με προσκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Μερίδα Ανάπτυξης και ήταν εκεί ο Λουί Επίσης, ο πρόεδρος της ε, Εθνοσυνέλευσης Μπουρκίνα Φάσο ήταν παρόν. Και τώρα κυρία Μπλάνκο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ναι, καλημέρα σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλ που είχατε αυτή την πρωτοβουλία της ε, διοργάνωσης αυτού του σεμιναρίου που πραγματικά είναι απολύτως αναγκαίο αυτή τη στιγμή της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ ειδικά την κυρία Μαρόκ που η δική της Ε, τον κύριο Μάνο, συγγνώμη, ε, που η παρουσίασή του μου φάνηκε πολύ καλή. Δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο του, κυρίου, του Manpower, τον κύριο Άρκλες. Και θα σας πω γιατί. Ε, στην παγκόσμια κρίση που είμαστε βυθισμένοι, οι λιγότερο ευνοημένες χώρες θα υποφέρουν τις επιπτώσεις της κρίσης υπό τη μορφή μιας κρίσης ε, στα τρόφιμα, επισητιστικής κρίσης. Ενώ άλλες ε, χώρες πλήττονται στον ε, χρηματοοικονομικό τομέα. Οι αναδιόμενες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η, και η Βραζιλία και όχι μόνο οι χώρες ΑΚΕ, αλλά και οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής θα πληγούν βαθύτατα από αυτή την κρίση εάν ενώσουμε κάτι το οποίο είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η συνεργασία για την ανάπτυξη, η, συνεκτικότητα στην πολιτική ανάπτυξη, ούτω ώστε να βοηθήσουμε την κατάρτιση των μεταναστευτικών ροών, την εκπαίδευση των μεταναστευτικών ροών, ούτω ώστε να μπορούν να διαβιούν σε αξιοπρεπείς και ανθρώπινες προϋποθέσεις, νομίζω ότι ε, θα ε, καταφέρουμε να εξέλθουμε από αυτή την ε, παγκόσμια κρίση. Και επιτρέψατε μου να σας πω στο τέλος και συγχωρέσατε μου που μακρηγορώ. Οι μετανάστευτες οι μετανάστες συγγνώμη, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην πλειοψηφία τους στη χώρα προέλευσης. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή ε, καταρτίζει προγράμματα επαναπατρισμού τα οποία δυστυχώς δεν επιφέρουν αποτελέσματα. Γιατί ε, στις χώρες αυτές τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από τα δικά μας. Ας μην είμαστε υποκριτές κυρίες και κύριοι, να δούμε κατάματα την αλήθεια. Το λόγο σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην κυρία Άννα Γκόμες από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει μια προαιώνια ιστορία εξαγωγής εργατικών χεριών και μια δεκαετή παράδοση εισαγωγής εργατικών χεριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταπολεμήσουμε την, το δημογραφικό πρόβλημα και για να εξισορροπήσουμε ε, τα ταμεία μας των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ζούμε μια παγκόσμια κρίση. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις και κανόνες σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που δεν το έχουμε. Θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Ντόισλερ. Δεδομένου δεδομένου του ρόλου των εμβασμάτων. Στη βοήθεια αυτών των χωρών, στις επενδύσεις προς αυτές τις χώρες. Και παρά τις εκκλήσεις που γίνονται στις ε, χώρες μέλη προκειμένου να σεβαστούν ε, τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να διευκολύνουμε τις ροές αυτές ε, από τα εμβάσματα και για να απαλύνουμε την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες κρίσης. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες που δεν σεβόταν τις αναπτυξιακές τους δεσμεύσεις όπως προλεβόταν από τον ΩΣΑ. Ε, σήμερα με την κρίση λοιπόν θα, θα τις σεβαστούν ακόμη περισσότερο. Θα δώσουμε λίγα λεπτά στους εισηγητές να απαντήσουν εφόσον τον το επιθυμούν. Ο κύριος Άκλες, εφόσον επιθυμεί από τη Manpower, να πάρει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι θαυμάσια αυτά τα ερωτήματα. Δεν μπορώ να απαντήσω λεπτομερώς. Θα ήθελα να εστιάσω στην ερώτηση αυτή, ότι δεν υπάρχει διεθνής φορέας υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση σε, αυτή την, όλο αυτό το σύστημα, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν υπάρχει, το χρειαζόμαστε. Μίλησα ε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ζήτησα ε, να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει ε, διάφορες οργανώσεις του ΟΗΕ να σκεφτούν, να συσκεφτούν από κοινού για να δουν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο φορέα. Εγώ τους τα είπα, αλλά βέβαια με αγνόησαν. Όσα θα συνεχίσει την προσπάθειά του, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την παγκόσμια αυτή ύφεση. Thank Uh, θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στις πολιτικές. Τα Υπουργεία Εξωτερικών, τα Υπουργεία Εργασίας και τα Υπουργεία Ανάπτυξης θα πρέπει να συνεργαστούν. Δεν υπάρχει αρκετό συντονισμός. Δεύτερον, έχω μεγάλες ανησυχίες ότι οι χώρες που είναι δωρήτριες δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία και η χρηματοδότηση της βοήθειας δεν είναι φιλανθρωπία, είναι πολιτικές επενδύσεις ε, για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Στις χώρες δωρήτριες η κοινή γνώμη θεωρεί ότι αυτό είναι απλώς υποστήριξη και απλώς βοήθεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερα επιχειρήματα για να πείσουμε το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι στρατηγικές επενδύσεις αυτές και σε καμία περίπτωση φιλανθρωπία. Είναι δύσκολο να τους πείσουμε όμως, λέει ο κύριος Μπορέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Αλλά από αυτά που άκουσα ε, σκιαγραφίσατε μια εικόνα μάλλον ζωφερή θα έλεγα. Σε ό,τι αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, η ανάπτυξη και η μετανάστευση είναι δύο από τους τομείς που πρέπει να κάνουμε προσπάθειες. Θα πρέπει να έχω μια παγκόσμια προσέγγιση για τη μετανάστευση και μια παγκόσμια, και μια παγκόσμια προσέγγιση για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε την ελαφρομετανάστευση, την νόμιμη μετανάστευση και τη μετανάστευση σε σχέση με την ε, ανάπτυξη. Αυτή η παγκόσμια προσπάθεια ε, υποσκάπτεται τώρα λόγω της κρίσης. Αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να την διατηρήσουμε την παγκόσμια προσέγγιση και να κάνουμε κάτι για την ε, παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Να μην στρεφόμαστε προς τα μέσα, να μην ομφαλοσκοπούμε ε, όλοι ομφαλοσκοπούμε, κάνουμε διάφορα σχέδια για την ανάκαμψη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα ήταν κίνδυνος αν ξεχάσουμε τις χώρε από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Και αυτός ε, είναι ο λόγος γιατί που ο πρόεδρος Μπαρόσο και η Κομισιόν δουλεύουν για να υπάρξει ένα εξωτερικό σχέδιο ανάκαμψης. Ε, για να πούμε ότι εμείς Ευρώπη δεν ξεχνάμε τον αντισόμενο κόσμου, θα διατηρήσουμε τι δεσμεύσει για την επίσημη αναπτυξιακή ανάπτυξη, θα βρούμε καινοτόμου τρόπου για να βοηθήσουμε τι χώρε τι αναπτυσσόμενε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στι αναπτυσσόμενε χώρε, να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση εκεί, που είναι προπόθεση για την κυκλική μετανάστευση, για την επιστροφή των μεταναστών και για πολλά άλλα πράγματα. Η απάντηση αυτή θα είναι η απάντηση της Κομισιόν. Θα υποστηρίξουμε και θα αναπτύξουμε μια παγκόσμια προσέγγιση. Θα κάνουμε κάτι για την παγκόσμια κρίση και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είστε προσκεκλημένοι στο μπουφέ εδώ έξω από την αίθουσα. Επειδή καθυστερήσαμε 10 λεπτά, ε, θα αρχίσουμε 10 λεπτά αργότερα. Παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ στις 2 και 10. Στις 2 για να ξεκινήσουμε μάλλον στις 2 και 10. The interpreters have to know that we'll start 10 minutes late. Thank you.